βάσει του άρθρου 137.2 του εσωτερικού κανονισμού. Έλαβα από την Επιτροπή ΕΝΒΗ το αίτημα για ε, διερευνητική γνωμοδότηση τη ε, ΕΟΚΕ για την υλοποίηση τη περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση στους τομείς όπου υπάρχουν ε, κενά. Δηλαδή την ατμοσφαιρική ρήπανση, τα ύδατα και τα απόβλητα. Εάν μέσα σε 24 ώρε καμία κοινοβουλευτική ομάδα ή ομάδα βουλευτών που φτάνει τον αριθμό ψήφων δεν προβάλλει αντίρρηση, θα θεωρηθεί εγκεκριμένο το θέμα και θα ψηφιστεί.